Okay, colleagues, I think we should make a start because it's a little bit later than planned. Καλημέρα σας και ξεκινούμε λίγο αργότερα από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Άρθρο 15, διαφθορμένος διάλογος, πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συναντήσαμε τον κύριο Στυλιανίδη. για να συζητήσουμε μαζί του βέβαια και το προγραμματισμό για το 19 που βέβαια θα έχει περιορισμένη έκταση λόγω εκλογών και εγκαθίδρυση της νέας επιτροπής, αν και δεν νομίζω ότι ε, θα έχουμε νέες προτάσεις, αλλά πολύ γρήγορα, αλλά ήταν καλή ευκαιρία να συστήσουμε με τον ε, Επίτροπο. Και να ακούσουμε τις απόψεις του για την προσεχή περίοδο, την προεκλογική. Αλλά βέβαια νομίζω έχει έρθει και η ώρα να κοιτάξουμε μια και κάποιοι από εσά θα ξανακλεγείτε, τι προτεραιότητες πρέπει να ορίσουμε για την προσεχή βουλευτική περίοδο. Πριν από λίγο ήταν, πριν από τη Μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση εδώ ο Επίτροπος, ε, πριν από μερικές εβδομάδες μόλις και συστήσαμε τα προγράμματα. Τον ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερος που ήρθε σήμερα. Ωστόσο, από την προηγούμενη του επίσκεψη δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Φαντάζομαι πολύ ενδιαφέρον το περίμεναν οι συνάδελφοι. Κάπου τον Ιούνιο περιμένουμε το νέο πρόγραμμα, τα νέα προγράμματα και ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει εάν η ανακοίνωση θα έρθει στην ώρα της. Είδαμε και με κυβερνητικές οργανώσεις, εκπροσώπησης πολιτών για το Πουδουπού. Ακούσαμε τις απόψει τους, μπορούμε να τις μεταφέρουμε και στον Επίτροπο. Κύριε Μιμίτσα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αξιότιμοι Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Από τις αρχές της ανάληψης εντολής της Επιτροπής σα. Ε, είχαμε μεγάλη συνεργασία και πρόοδο στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια βασικά σημεία πρόοδου στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Καταρχάς, το φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο και θεματολόγιο 2030 της ε, Οργάνωσης των Εθνών για την εκρίζωση της φτώχειας και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης συμφωνήθηκε με μια κοινή ευρωπαϊκή συνένεση που συνοδεύει το θεματολόγιο αυτό και μεταφράζει το θεματολόγιο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των στόχων του. Επίσης είχαμε και ένα φιλόδοξο ε, σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων για την υποστήριξη των στόχων μας ως προς την αναπτυξιακή πολιτική. Άνευ προηγουμένου ε, μεγάλη πρωτοβουλία σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για την ε, για τον τερματισμό της βίας βάρος γυναικών και κοριτσιών που είναι εν εξελίξη. Βεβαίως πολλή δουλειά ακόμα μένει να γίνει στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο και έτσι την εισήγησή μου θα την εστιάσω στις κύριες προτεραιότητες που ακόμη επιδιώκουμε. Ε, πρώτον, νέε συμφωνίε εταιρικής σχέσης μετά ή διευθετήσεις μετά το Κοτονού. Κοινές προτεραιότητες με τους εταίρους μας από την ΑΚΕ. Έχουμε συζητήσει και προσδιορίσει με πολλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα με την ε, υποστήριξη του κυρίου Νόιζα. Ε, απόφαση του Συμβουλίου και εντολή υπουργική από τους εταίρους ΑΚΕ αναμένεται σύντομα έτσι ώστε να δοθεί εντολή για την εκκίνηση των τυπικών διαπραγματεύσεων πριν από τον Αύγουστο. Θεωρώ ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ Επιτροπής Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, για το όλο πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων και των ε, γενικών εταιρικών σχέσεων ε, και συμφωνιών. Ωστόσο, χρειάζεται να εξευρεθεί σε για ορισμένους τομείς συμφωνία με τα κράτη-μέλη για το μέλλον της συμφωνίας, τη διάρκεια της και το μεταναστευτικό. Ανησυχίε που ορισμένοι από εσά έχουν εκφράσει με υποχρεώνω να σα διαβεβαιώσω ότι μέρος της διαδικασία αυτής και των διαπραγματεύσεων ε, αποδεικνύουν την προσήλωσή μας στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης αλλά και την ε, ε, ευρύτητα πολυτομεακών εταίρων με τους οποίους συνομιλούμε σε διάφορα επίπεδα. Δεύτερο, στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμερική, πάλι κομμάτι του προγράμματο εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ ετοιμάζουμε μια σειρά από περιφερειακέ στρατηγικέ που θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν με τον ίδιο τρόπο μια ευρεία προσέγγιση για τι κοινέ ε, εταιρικέ σχέσει για τις ευρωπαϊκές ε, εταιρικές σχέσεις και κοινέ προτεραιότητες σε συνεργασία με τις χώρες Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβική. Περιμένουμε να είναι έτοιμο τον Αύγουστο, το φθινόπωρο για να σας το παρουσιάσουμε. Με βάση βέβαια το θεματολόγιο 2020, τη δουλειά που έχουμε κάνει με την εταιρική σχέση ΑΚΕ και εδώ μπορούμε να προσδιορίσουμε πέραν άλλων ζητημάτων στις στρατηγικές σε σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και ένα σαφές όραμα για την συνεργασία με χώρες υψηλού επίπεδου ανάπτυξης και άρα εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως ανισότητες και την ανάγκη ανοικοδόμησης κοινωνιών και οικονομίων οι οποίες προσανατολίζονται προς την βιωσιμότητα αλλά και ταυτόχρονα μεγιστοποίηση για τις αναδυόμενες, νέες αναδυόμενες οικονομίες με βάση τα κοινά μας συμφερόντα και αξίες. Πρέπει να προσδιορίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για μεγιστοποίηση των αμοιβαίων ωφελημάτων αυτής της συνεργασίας ε, με αδελφοποίηση, τριμερείς συνεργασίες, ενίσχυση άλλων μορφών συνεργασία και να κοιτάξουμε και πού αλλού μπορούμε να επαναλάβουμε αυτές τις μορφές συνεργασίας. Βεβαίως όχι εις βάρος της δουλειάς που αλλου μπορουμε να επαναλαβουμε αυτες τις μορφες συνεργασια βεβαιως οχι εις βαρος της δουλειας που κανουμε σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Τρίτο θέμα, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασύνδεση με την ε, μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. έχουμε να ετοιμάσουμε μια νέα στρατηγική συνδεσιμότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας ε, μέχρι το φθινόπωρο. Βέβαια η συνδεσιμότητα έχει πολύ μεγάλο δυναμικό και για την υλοποίηση του θεματολογίου 2020 και γενικά για την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, μεταφορές, εμπόριο, ενέργεια, ψηφιακές υπηρεσίες, ε, ε, διαπροσωπικές επαφές είναι κομμάτι, είναι κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και τη συνδεσιμότητα στόχο έχει να εξασφαλίσει ότι δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο. Επίσης, η συνδεσιμότητα σημαίνει ότι θα συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους εταίρους μας στην Ασία. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει την, ε, τις επαφές με τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης περιοχής ε, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ιαπωνίας, ταυτόχρονα όμως προβάλλοντας και προάγοντας την πολυμερή συνεργασία, κυρίως μέσω τη ΑΣΕΑΝ με διάφορες χώρες της περιφέρειας. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του προγράμματο εργασία βεβαίω ήταν η συνεργασία ευρωπαικη Ευρωπαϊκή Ινδίας και εδώ επιδιώκουμε συνεργασίε με πιο προηγμένε χώρε μεταξύ των οποίων βεβαίω η Ινδία, ε, χώρες που έχουν κοινέ αξίε και στόχου με μας. Η νέα στρατηγική στρατηγική Ευρωπαϊκή Ινδία θα εστιαστεί στου τρει πυλώνες ε, του παγκόσμια τάξη με βάση το κράτο δικαίου και βιώσιμη ανάπτυξη, διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ενίσχυση τη αμοιβαία ευημερία και κατανόηση. Και Γνωρίζω βέβαια ότι έχει έρθει η ώρα να κοιτάξουμε το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και επιτρέψτε μου γι' αυτό λόγο να σας πω και γι' αυτό δύο λόγια. Προτάσεις δηλαδή του Πουδουπού που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Μαΐου. οι εξειδικευμένε τομεακέ προτάσει θα κατεθούν μόνο 14 Ιουνίου και θα υπάρχουν κάποια μόνο συγκεκριμένα και περιορισμένα μηνύματα σε σχέση με την εξωτερική δράση και αναπτυξιακή βοήθεια. Καταρχά, ε, πρόκειται για ένα κλάδο που χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως ως το χώρος ε, προτεραιότητας για το μέλλον δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ιδιαίτερο συμφέρον δηλαδή να αναλάβουμε δράση και να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στον χώρο της αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας και οι δαπάνες στο πεδίο αυτό δεν θα πρέπει να περιοριστούν, δεν θα πρέπει να υποστούν πλήγμα λόγω του εις του Ρωμανού Βασιλείου και των συναφών συνεισφορών στον προϋπολογισμό. Οι δαπάνες λοιπόν για την εξωτερική δράση θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά και πέραν των τωρινών επιπέδων. 133 δισεκατομμύρια για εξωτερικές δράσεις. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο θα γνωρίσει αύξηση του 26%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μερίδιο που έχει στη συλλογική προσήλωση τη συλλογική αλλά και την επιμέρους των κρατών μελών για την ε, αύξηση κατά 0,1 επί του ΑΕΠ της ε, αναπτυξιακής βοήθειας οπωσδήποτε θα την τιμήσει με τον τρόπο αυτό. Οι συνολικές λοιπόν δαπάνες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την εξωτερική δράση θα πρέπει να πληρούν ε, τα κριτήρια της αναπτυξιακής βοήθειας σε κάθε τομέα με ένα 95% των συνολικών εξωτερικών δράσεων στην κατηγορία ODA. Και έτσι βέβαια θα τις ε, καταγράφουμε και στο μέλλον τις δαπάνες αυτές. Ε, επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία ε, οργάνωση των μέσων εξωτερικής δράσης πέραν των θεματικών ή γεωγραφικών μέσων προτείνουμε και ένα ευρύτερο μέσο για την ανάπτυξη της γειτονίας και τη διεθνή συνεργασία με ένα φάσμα οικουμενικό, παγκόσμιο, αναγκαίο και συναφές με την έννοια της οικουμενικής ε, Εφαρμογή του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 21ου αιώνα και του στόχου τη χιλιετία. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συνολικά την ενίσχυση και της εποπτεία και των δημοσιονομικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προκείμενη περίπτωση, Όπω πολύ σωστά ε, ε, και επιμακρών έχει απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνεται η, ανάπτυξη, η αύξηση του αναπτυξιακού ταμείου με βάση και τη λογική της καλύτερης οργάνωσης και χρήσης των πόρων μας, η οποία θα πρέπει να ε, βαίνει παράλληλα και προς την εξασφάλιση ευελιξίας μέσα από τον προϋπολογισμό, παραδείγματι δυνατότητα επανε... επαναγραφής κονδυλίων όταν χρειάζεται. Και αυτό προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και βέβαια να στηριχτούν εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθεια αυτή στις χώρες εταίρους. Ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να περιορίσει την επιβάρυνση για τους χώρες εταίρους και τους λοιπούς συνεργαζόμενους όπως οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών αλλά ταυτόχρονα και την ευρωπαϊκή πλευρά των υπηρεσιών, των φόρτων για τις υπηρεσίες που έχουν την εποπτεία και την παρακολούθηση. Έτσι λοιπόν οι ιδιαιτερότητες εξωτερικών ε, πολιτικών θα διατηρηθούν βέβαια ε, και θέλω να καταστήσω σαφές ότι ένα εργαλείο, ένα μέσο ε, ευρεία εφαρμογή δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μόνο μία πολιτική. Αντιθέτως, έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε ακόμη περισσότερο τις πολιτικές μας επιλογές και αυτό το μέσο, το αναπτυξιακό, να τεθεί στην υπηρεσία αυτή της πολιτική και με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση που στόχο έχει κατά κύριο λόγο την εκρίζωση της φτώχειας ε, μπορούμε να έχουμε και την ε, ορατότητα, την ε, προβλεψιμότητα, την έννοια της ιδιοκτησίας για τις χώρες εταίρους και τους λοιπούς άλλους παράγοντες και χαρακτηριστικά της συνεργασίας πάντα στο προσκήνιο. Βεβαίως και εμείς θα είμαστε καλύτερα σε θέση για μια εις βάθος ανταλλαγή απόψεων κατά τη στιγμή της υιοθέτησης της νομοθετικής πρωτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο σε ένα μήνα περίπου. Και βέβαια περιμένω τις δικές σας προτάσεις και τις ε, φιλόδοξες προτάσεις ιδιαίτερως και απαιτήσεις έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι ε, φιλοδοξίες μας και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου προσφέρατε για διαρθρωμένο διάλογο και για συμβολή στη συνεργασία ε, εν βέβαια και του προγράμματος εργασίας αλλά και του προσεχού σπουδού. Ευχαριστώ. Καλώς ευχαριστούμε για την εισηγησή σας κύριε Επίτροπε. Βλέπουμε ότι διατηρείται το ενδιαφέρον σας και το ρυθμό των εργασιών. Ποιος θέλει το λόγο. Νόιμπερτ. Για πες μας να ξέρουμε πόσοι θέλουν να, λάβουν το λόγο. Μπόγκτεν, εσύ πρώτος. Βέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Επίτροπε που ήρθατε να μας δείτε. Παρατηρήσεις και ερωτήσεις από πλευρά της δικής μας πολιτικής ομάδας όσον αφορά το θεματολογειο 2020-30 και τους ε, βιώσιμους εμτσέκους στόχους. Έχουμε αυτή την γνωμοδότηση για τη σχέση μας με την Αφρική. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σημαντική προσπάθεια να γεφυρωθούν οι ανισότητες και να αντιμετωπιστούν οι δεσμενείς διακρίσεις και θα πρέπει να διατηρήσουμε τις προσπάθειές μας. Τι θα κάνετε τόσο ώστε να έχουμε ε, την υλοποίηση αυτών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και πέστε μας Δύο λόγια γι' αυτό. Επίσης, με τον Όρμπρετ είμαστε συνεισηγητές για το θέμα της συνένεσης για την ανάπτυξη. Και αυτό το θέμα έχει σχέση με το θεματολογιο 2030 και υπάρχει κάτι το οποίο ακόμη εκκρεμεί όσον αφορά το ε, πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη. Εσείς Πρόκειται να καταρτήσετε κάποιο σχέδιο πριν το τέλος της θητείας. Νόιζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εισήγηση, η οποία καταγράφει τα... Ε, μάλλον τα, τα βασικά στοιχεία μας τα περιέγραψε ο Μπόγκταμ για την στένεση για τις ε, χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Θα ήθελα να φέρω ένα νέο σημείο ωστόσο, γιατί περιμένουμε το φθινόπωρο ε, να προχωρήσουν και οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΑΚΕ και τις δικές μας βέβαια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη συνέχεια που θα δοθεί στην φάση μετά το Κοτονού. <coughs> Βεβαίως έχουμε δώσει με την εμπιστοσύνη μας εντολή διαπραγματευτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε ως Κοινοβούλιο να ενημερωνόμαστε. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια καλή λύση. Για το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, Νομίζω ότι είναι κάπως ε, διαφιλονικούμενο τουλάχιστον στα κράτη-μέλη εάν ε, θα οριστούν 20-25 χρόνια για να απλώς θα δοθεί μια παράταση της ε, προηγούμενης συμφωνίας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διευκρινιστεί. Σημασία έχει για μένα βεβαίως τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη. να εγκαταλείψουμε πλέον στη συζήτηση για την αναπτυξιακή συνεργασία την προσήλωση ορισμένων ορισμένων κρατών μελών στη συζήτηση μόνο στο μεταναστευτικό. Γιατί βεβαίω ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι τη αναπτυξιακή βοήθεια στο μεταναστευτικό, αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Δεν εξατλείται εκεί το θέμα. Και βεβαίω υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν ε, δώσει όλη τους την προσοχή μόνο στη μετανάστευση, αλλά σε αυτό θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε ώστε να αλλάξει η εστίαση. Και αν κοιτάξουμε τη συστηματική ε, διάρθρωση των νέων προτάσεων με την έμφαση που βλέπουμε να δίνεται στην μετανάστευση, αυτό να αποτελεί και μια παραχώρηση προς τα κράτη-μέλη, ώστε τα κράτη-μέλη να αισθανθούν την ικανοποίηση ότι, ικανοποίηση ότι έχει όντως δώσει ε, την ε, δέουσα σημασία στη μετανάστευση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά υπογραμμίζω η αναπτυξιακή συνεργασία έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να την ε, εξαντλήσουμε σε αυτό. Επίσης για τα θέματα ΑΚΕ και τους περιφερειακούς πυλώνες, ε, χώρες Καραϊβικής, Λατινική, Αμερική, πάνε μαζί ή χώρες του Ειρηνικού υπολογίζονται στην Ασία και ίσως χάνονται κάπως ε, οι χώρες του Ειρηνικού, δεν τους δίνουμε αρκετή σημασία δηλαδή μέσα σε αυτή την ε, γεωγραφική ταξινόμηση. Μήπως λοιπόν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη, κάποιος σχεδιασμός για μια ξεχωριστή αντιμετώπιση των χωρών της Καρυβικής αφενός και του Ειρηνικού αφετέρου, φερρυπίν με χωριστά πρωτόκολλα, γιατί χρειάζεται και δυνατότητα προγραμματισμού και πάνω απ' όλα μεσοπρόθεσμα προγράμματα να έχουμε και νομίζω ότι η δυνατότητα της ευελιξίας μπορεί όντως να έχει μεγάλη χρησιμότητα όταν εφαρμόζεται σε πραγματικούς χρόνους, αλλά πάλι χρειάζεται να έχουμε μια προβλεψιμότητα στις ε, μεσοπρόθεσμες λύσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Χόιπρο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα. Πιστεύω ότι Πολλά από αυτά που θα ακούσετε σήμερα ήδη τα γνωρίζατε. Πρέπει δυστυχώς ε, να πούμε τα γνωρίζετε γιατί είναι πολύ το ο που δεν έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος και πάντα αναγκαζόμαστε να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες απαιτήσει. Επί παραδείγματι, απέτηση για νομοθετική πρωτοβουλία για, ε, προϋπο... για πρότυπα παραγωγής στην κλωστοϊφαντουργία ή για την ε, για τις συνέπειες σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες σε αναπτυσσόμενα κράτη παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ε, παράδειγμα της αρπαγής γης είναι ένα από αυτά τα οποία μας απασχολούν και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων και των θυμάτων και όχι των επιχειρήσεων όπως κάνει τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω και μια νέα πρόταση, ελπίζοντας ότι θα εγγραφεί στο πρόγραμμα εργασίας και θα περιληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια προσέγγιση, υποτίθεται, με εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αναπτυξιακή τη βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά όπως είπα έχουμε πολύ συχνά παραβιάσει των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μέσα σε έργα και σχέδια της αναπτυξιακή βοήθειας που δεν μπορούμε πάντα εξ ολοκλήρου να αποφύγουμε ή να αποτρέψουμε. Και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα, το, σχέδιο της, το έργο που έχουμε στην Κένια, Μπάρτερ, θα ήταν καλό να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά. Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ή θα πρέπει καλύτερα να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, προσφυγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε οι πολίτες οι οποίοι μέσα σε σχέδια υποστηριζόμενα από την αναπτυξιακή μας βοήθεια ε, να έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση παραβιάσεων να προσφεύγουν. Βεβαίω θα είναι διοικητικέ οι προσφυγέ, διοικητικό ο μηχανισμό. Πρέπει να υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία ώστε ένα θύμα να μπορεί να έχει τη δυνατότητα πρώιμα να καταθέτει σε πρώιμο στάδιο, να μπορεί να καταθέτει και μάλιστα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις, ε, ε, τα παράπονά του, τις ενστάσεις του, έτσι ώστε να μην ε, κλιμακώνεται η κατάσταση όπως είδαμε να συμβαίνει λόγω των καθυστερήσεων στην Κένια. Και βεβαίως αυτός ο μηχανισμός των προσφυγών πρέπει να είναι διοικητικός, έτσι ώστε να, να, λειτουργεί και ως προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας άσκησης των ένδικων ε, ε, μέσων και βοηθημάτων. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ήδη έχετε δεχθεί. Και θα ήθελα επίσης να, να προσθέσω μετά τα, είπαν, μετά τα όσα είπαν οι συνάδελφοι Βέντα και Νόιζερ ότι πρέπει και το έχουμε ήδη σημειώσει στη συνένεση, να υποστηρίξουμε περισσότερο τις ε, ε, περιβαλλοντικές γεωργικές μεθόδους. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό σε επίπεδο Εθνούς Γεωργίας και Τροφίμων. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς εδώ με βάση τα πρότυπα αυτά και έχουμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο τώρα το οποίο θα ήταν σκόπιμο στο χώρο αυτό να δώσει επαρκή μέσα. Γιατί λέμε ότι θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στην οικολογική γεωργία και θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Γεωργίας και Τροφίμων, αλλά βλέπω να, είμαστε, να υπολοιπόμαστε πολύ και πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Just take answers to those first απαντήστε σε αυτούς τους τρεις και θα κάνουμε άλλον έναν γύρο ερώτα απαντήσεων. Κατόπιν, Ελίς Λάιν. Ρούμπιχ και Σαργεντίνη. Αυτή είναι στον δεύτερο γύρο. Αλλά ας κάνουμε πρώτα τον πρώτο γύρο. Uh, the implementation η υλοποίηση αυτών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης SDG είναι ο βασικός άξονας της πολιτικής μας. Ήταν και θα είναι την επόμενη περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει δραστηριότητα και είναι σημαντικός παίκτης και φιλόδοξος όσον αφορά την κατάρτιση του θεματολογίου για αυτούς τους στόχους SDG. Θα πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα, να συνεχίσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των στόχων για όλο τον κόσμο σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους μας αλλά και στο εσωτερικό της Ένωσης. Βέβαια έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα πάρα πολύ σημαντικό αυτή η στόχη. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν παντού κάτι το οποίο για μας προϋποθέτει συνδυασμό διαφορετικών πολιτικών προϋποθέτει δράσεις που θα έχουν μεταξύ τους συνεκτικότητα και συνέπεια. Αυτές οι δράσεις θα έχουν μπούσουλα αυτή την νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση. Αυτό θα μας κατευθύνει. Επίσης, θέλουμε όμως όλα αυτά να γίνουν συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα έργα για κάθε χώρα εταίρο μας. Και θα συνεργαστούμε φυσικά και με το Κοινοβούλιο, θα έχουμε και τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση όπου και εκεί θα εμπλακεί το κοινοβούλιο τώρα. Θα πρέπει να καθορίσουμε τα συγκεκριμένα μέσα πολιτικής, τους τρόπους υλοποίησης αυτών των SDG, και θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η πολιτική θα ασκηθεί και σε περιφερειακό επίπεδο. πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει μετά την Κοτονού. Να δούμε πώς μπορεί να συμβαλεί η Ευρώπη για αυτούς τους στόχους. Τέλος, το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο και οι σχετικές προτάσεις θα είναι στόχοι κοινή. Στο μέλλον και ελπίζουμε αυτή η περίοδο να γίνεται πιο σύντομη, οπότε και θα δούμε με τι μέσα θα κινηθούμε σε έναν νομοθετικό πλαίσιο για να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των SDG. Η συνένεση για την ανάπτυξη αποτελεί ένα έγγραφο που είναι η πηξίδα για το σύνολο του έργου μας, οπότε Αυτό θα μας καθοδηγήσει όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο αυτής της συνένεσης. Θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι και όσο γίνεται πιο ξεκάθαροι. Να δούμε πώς στην επόμενη φάση θα περάσουμε κάποια διαπραγμάτευση και θα έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την ε, υλοποίηση αυτής της ε, συνένεσης πάντως. Σήμερα δεν προβλέπω κάποιο τέτοιο πρόγραμμα δράσης. Θα πρέπει να γίνει πάντως συνένεση πράξη. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμό. Σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Συμφωνώ επίσης. 100% ότι η όλη η αναπτυξιακή πολιτική μας θα πρέπει να καλύψει και άλλους τομείς και άλλα θέματα και στόχους που σχετίζονται άρκετα με την ανάπτυξη, όπως ας πούμε η μετανάστευση. Θα πρέπει όμως να δούμε απομονωμένα την μετανάστευση σαν κάτι ξεχωριστό ως στόχο της αντιξιακής πολιτικής. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη σε σχέση με τις αιτίε της μετανάστευσης. Άρα ε, το θέμα είναι η κρίζωση της στόχιας και αυτό είναι ε, ο σύνδεσμος το ΣΥΠΗΝ μεταξύ ανάπτυξης και μετανάστευσης. Τα προγράμματα, τα μέτρα κατά της φτώχειας συγκεκριμενοποιούν αυτή τη στενή σχέση μετανάστευσης με ανάπτυξη. Δεν χρειαζόμαστε ξεχωριστό μέσο πολιτικής για την μετανάστευση. Τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι ο καλύτερος τρόπος τόσο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις αιτίες της μετανάστευσης, δηλαδή να βελτιώσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις χώρες που είναι εταίροι μας. Κάποια άλλα θεματάκια υπάρχουν για την περίοδο που θα ακολουθήσει την Κοτονού ζητήματα με τους εταίρους μας τη Οπότε, όλα αυτά ελπίζω επιτυχώς να διεκπαιριωθούν και να ρυθμιστούν τις αμέσωπες εβδομάδες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η διαπραγματευτική εντολή της Ένωσης. Αυτό θα γίνει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Οπότε είμαστε έτοιμοι για τις δημοτεύσεις με τους εταίρους και; Και να πάμε σε μια σφαιρική συμφωνία για το μέλλον και να δούμε τα επιμέρους περιφερειακά πρωτόκολλα ή επιμέρους συμφωνίες. Τώρα για την αρπαγή των γεών, για διάφορα επιμέρους θέματα όπως η γεωργία, όπως η ιατροφική ασφάλεια. Για τα σχετικά προγράμματα είμαστε έτοιμοι. Να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτωπα με πάσα αναπτυξιακή μας δράση. Επίση να αναβαθμίσουμε την προσέγγιση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη συνεργασία μας. Να υπάρχει συγκεκριμένη σχέση μεταξύ ανοιξέγων δράσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βαθμό του δυνατού. Οπότε, προσβλέπω στη συνεργασία με τα κοινοβούλια, όποτε επιβάλλεται. Οπότε, λέγω θέλουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής μας της προσέγγισης να έχουμε η αξιολόγηση επιπτώσεων για την πρωτοβουλία μας. Κάτι το οποίο θα μας πάει στην επόμενη φάση πρωτοβουλειών. Ε, αυτό θα γίνει βέβαια σε αυτή την εντολή, αλλά μετά. Οπότε να συνεχίσουμε σε ε, αυτή την ρότα του διαρθρωμένου διαλόγου για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να είναι αποτελεσματική η αναπτυξιακή μας πολιτική η πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, ζητήσω συγγνώμη γιατί άργησα. Ε, ζητούσαμε τη Σεσίλια Μάλστρομ για διάφορα θέματα σχετικά με το εμπόριο. Όπως γνωρίζετε, ε, συνδέεται αυτό το θέμα με την αναπτυξιακή πολιτική και την αντιμετώπιση των στόχων από τη μία τη φτώχεια και από την άλλη η βελτίωση των εξαγωγών και πώς θα μπορούσαμε να ε, επιτύχουμε μια δίκαιη πολιτική και στους δύο τομείς ε, με συμβολή ε, στο διεθνές εμπόριο και στην ανάπτυξη. Όλα αυτά μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν άμεση σχέση με τη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από τη μία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες ζητούν περισσότερες πηγές ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιολογικών ε, καυσίμων στο τομέα της ενέργειας και ταυτόχρονα ε, γίνονται πολλές εισαγωγές φοινικέλεου. Και τώρα κινούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση και Προσπαθούμε να ε, απαγορέψουμε το φινικέλαιο. Φυσικά υπάρχουν χώρες όπου μικροί γεωργοί εξαρτώνται από την παραγωγή ε, φινικέλαιου και τέτοιες αποφάσεις για αυτούς είναι σκέτη καταστροφή. Και έχω την εντύπωση ότι η συνεργασία εντός της Επιτροπής πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί φυσικά υπάρχει σύγκρουση συμβερόντων ε, ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής. Οι ε, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 2 και 7 θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αντιφατικά, γιατί ο 2 αφορά την ασφαλή γεωργία και ε, ο στόχος 7 αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει λίγο, λοιπόν, ε, ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο αυτούς στόχους. Και πρέπει να ε, φροντίσουμε να λειτουργήσουμε προς το συμφέρον του, προστατεύοντας το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα προστατεύσουμε και τα συμφέροντα χωρών όπως η Μαλαισία που εξαρτώνται από την παραγωγή φινικέλου. και... γιατί αν δεν μπορούν να εξάγουν πια σημαίνει ότι εμείς πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες ή να κάνουμε νέες επενδύσεις εκεί για να τους προσφέρουμε εναλλακτικέ λύσεις και έχω την εντύπωση ότι έχουμε ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο να, για την εξάλληψη της ε, φτώχειας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας γιατί κάποιοι στο τομέα της ενέργειας πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για μας να αλλάξει η στρατηγική μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Ε, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει ε, τρόπος να αλλάξουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, Έλλη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε να μας κάνετε αυτή την παρουσίαση ενός συνολικού οράματος και βέβαια των αποτελεσμάτων που έχουμε εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και των ε, περαιτέρω βημάτων για την ε, αναπτυξιακή μας στρατηγική πολύ σύντομα τις εξής τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, θέλω να εκδηλώσω την προσδοκία μου για μια πιο συνολική πρόταση που περιμένουμε να δούμε στα τέλη Ιουνίου. Αυτά που έχουμε μέχρι τώρα διαβάσει, τώρα το Μάιο βεβαίως και είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά μένουν και κάποια σημεία ασάφεια σε σχέση με το ενιαίο αυτό μέσο. Και βεβαίως είναι πολύ λογικό να εξορθολογιστούν τα υφιστάμενα μέσα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των ε, γνήσιων στόχων της ε, ανάπτυξης και βέβαια της διαφάνειας και του δικαιώματος του Κοινοβουλίου μας να έχει μια εποπτεία της χρηματοδότησης που χορηγείται. Ε, δεύτερον, και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τάση ε, μέσα που κανονικά προορίζονται για την ανάπτυξη να αξιοποιούνται και για άλλους στόχους που δεν είναι άμεσα συναφείς με την ανάπτυξη, όπως, με, όπως σε παραδείγμα τον έλεγχο των συνόρων ή ανάπτυξη άλλων ε, δυνατοτήτων, άρα όχι καθαρά αναπτυξιακών στόχων και αυτό μας ανησυχεί. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε την τάση αυτή και πρέπει να δούμε και αυτό το ενιαίο μέσο πώς θα μας επιτρέψει να ε, παρακολουθούμε την ε, σωστή στόχευση των μέσων. Το accountability όπως λέμε. Και βεβαίως και με τη χθεσινή μας συνάντηση με τον Επίτροπο Στυλιανίδη είδαμε ξεκάθαρα ότι είναι πολύ μεγάλες ακόμα οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να υλοποιήσουμε τις διεθνείς μας δεσμεύσεις, αυτά που έχουμε συμφωνήσει για το 2030 με τις συμφωνίες των Παρισιών, των Παρισιών και όλα αυτά τα άλλα που και κανείς αυτό θα μπορεί σε τελευταία ανάλυση να υλοποιήσει και γι' αυτό η έκκληση προς εσάς και προς τα κράτη-μέλη για μια σαφή πολιτική βούληση που πρέπει να εκδηλωθεί προς τους στόχους αυτούς αλλά ταυτόχρονα συνοδεύεται και από τους απαραίτητους πόρους γιατί πολλές δεσμεύσεις λαμβάνονται επί χάρτου αλλά δεν υπάρχουν οι πόροι που απαιτούνται για να τις υλοποιήσουν. Και μια τελευταία παρατήρηση για την ε, αποστολή που πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγκάντα με την Επιτροπή μας. Όπως ξέρετε στην Ουγκάντα έχουμε 1.300.000-400.000 πρόσφυγες που βέβαια είναι πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων ε, και σε ε, σχέση με την επιβάρηση για τη χώρα αυτή, η οποία έδειξε μια πολύ προοδευτική στάση, κρατώντας ανοιχτές ε, τις συνοριακές της πύλες. Έφτασε μάλιστα μέχρι να τους δίνει από ένα μικρό κλήρο που μπορούν αμέσως να αρχίζουν να καλλιεργούν. Ίσως λοιπόν έτσι σε, μερικά χρόνια μπορούν να φτάσουν σε μια αυτονομία ως προς την εξασφάλιση του προστοζήν. Βεβαίως ε, εξήραμε την υποστήριξη από τις τοπικές ε, κοινωνίες ε, της υποδοχής και προσφοράς προς τους πρόσφυγες, κυρίως από τον Νότιο Σουδάν. Και αυτό γιατί Ξέρουμε ότι ε, και γι' αυτό επιμένουμε τα μέσα όλα που θα διατεθούν να ε, κατευθυνθούν κατευθείαν προ τους πρόσφυγε και τι τοπικέ κοινωνίε. Γιατί ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα κράτο με πολύ περιορισμένου πόρου και για κοινωνία με πολύ περιορισμένου πόρου. Και θα ήθελα ε, για το θέμα αυτό να πω ότι επισκεφθήκαμε μια σειρά από έργα της ΔΕΦΚΟ, της ΕΚΟ, του, του καταπιστεύματος για την Αφρική, έργα σημαντικά που μπορεί να αλλάξουν ε, ζωές ε, ανθρώπων, ε, να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση πόρων, στην επένδυση σε μικρές οικονομικές δραστηριότητες, σε εκτροφή ζώων και άλλες αντίστοιχες, σε πρακτικούς όρους δηλαδή και είδαμε ότι οι άνθρωποι μας που είναι εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ωστόσο η κρίση δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση ακόμα. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη στήριξη πάνω από όλα στους τομείς της ε, υγείας, υγειονομικής περιθάλψης, της εκπαίδευσης και κυρίως της δευτεροβάθμιας και χθε η ακόμη Επίτροπος επεσήμανε ότι είδαμε σχολεία με 2.000 παιδιά. Τάξεις με πάνω από 100 παιδιά η καθεμία. Αδύνατο να προσφερθεί ε, εκπαίδευση ποιοτική σε τέτοιου είδους συνθήκες. Και επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε εν τέλει ότι αυτή η κρίση θα μπορούσε να επιδεινωθεί κιόλα. Διότι έχουμε στην άμεση γειτονία το Νότιο Σουδάν με τραγικές συνθήκες, το Μπουρούντι, όπου δυστυχώς πολλές ανησυχίες ε, μας γεννούν οι εξελίξεις και ακόμα και το Κονγκό. Με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη καταφτάσει στην Ουγγάντα με στην πρώτη στο πρώτο κομμάτι του χρόνου, στις αρχές του χρόνου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αποστρέψουμε το βλέμμα, πρέπει να φροντίσουμε αυτοί οι πρόσφυγες να μπορούν να ξεφύγουν από τους καταβλισμούς και να μεταβούν σε αστικά κέντρα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή ακόμη για ενσωμάτωσή τους σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο που προσφέρεται και χάρη στη συνεργασία που προέκυψε από τη Συνοδοκορυφή της Νέας Υόρκης. Ευχαριστώ. Σάρχεν, τι και μετά Κέντζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας άκουσα και ε, η αλήθεια είναι ότι έχω την εντύπωση ότι προσπαθείτε να ε, τετραγωνίσετε το κύκλο. Ένας προπολογισμό δεν ε, είναι συνώνυμο μίας πολιτικής. Είστε επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη. Σημαίνει ότι κύρια προτεραιότητά σας είναι η εξάλληψη της έσχατης φτώχειας. Στη πολιτική Πώς ελέγχεις τις δράσεις μέσω του προϋπολογισμού. Πώς ελέγχεις τις δαπάνες ως βουλευτής, ελέγχεις τον προϋπολογισμό. Εμείς έχουμε το ε, δικαίωμα να ελέγξουμε τον προϋπολογισμό με έναν ενιαίο προϋπολογισμό είναι δύσκολο να ελεγχθεί μια πολιτική και να δούμε αν κινούμαστε προς την εξάλληψη της έσχατης ε, φτώχειας ή αν η αναπτυξιακή συνεργασία θα, χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Και σχετικά με την ευελιξία, αν γίνει κάποιο σεισμός κάπου, η ευελιξία είναι πρωταρχική σημασία, αλλά για την βιώσιμη εξάλληψη της έσχατης φτώχειας η ευελιξία είναι είναι κάτι πολύ κακό. Σκεφτείτε το ε, ε, ε, παράδειγμα που σας δόθηκε στην Ουγκάντα. Αυτοί οι πρόσφυγες από το νότιο Σουδάν θα μείνουν εκεί. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το Καταπαιδευματικό Ταμείο για την Αφρική που έχει διάρκεια δύο χρόνια. Αυτή η ευελιξία οδηγεί σε ανασφάλεια. Η ε, ευελιξία στο τομέα της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη σημαίνει περισσότερο κίνδυνο να χρηματοδοτήσουμε ε, δράσεις ειδικού σκοπού, αλλά όχι απαραίτητα για την υπεράσπιση των συμφερόντων χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα φτώχειας. Η εξάλληψη της φτώχειας χρειάζεται μακροπρόθεσμη δράση τα αποτελέσματα δεν θα είναι άμεσα. Η ευελιξία στον προϋπολογισμό είναι ό,τι χειρότερο για την αναπτυξιακή συνεργασία και θα ήθελα να καταλάβω στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πώς θα επιτύχουμε το στόχο του 0,7%. Δεν το βλέπω πιθανό και πώς εκ των προτέρων θα αποφασίσουμε ποιο κομμάτι του προϋπολογισμού ε, είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση δράσεων αναπτυξιακής βοήθειας. Πώς θα ξέρουμε πού έχουν δαπανηθεί τα χρήματα εκ των υστέρων, δεν μπορούμε να ξέρουμε, ε, ε, να ελέγξουμε κατάλληλα τις δράσεις. Και κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε, ε, μιλήσατε για την ανάγκη να υπάρξει ένα ε, διαφορετικό ε, χρηματοδοτικό εργαλείο για την μετανάστευση και μετά είπατε ότι η μετανάστευση πρέπει να είναι προτεραιότητα. Είπατε και κάτι διαφορετικά. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι όταν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη σε μια πολύ φτωχή χώρα, η μετανάστευση αυξάνεται. Και πάλι ε, πρόκειται για θέμα ε, γενιών. Αν ε, αναζητούμε άμεσες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του μεταναστευτικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν θα δαπανίσουμε τα χρήματα εκεί που πρέπει ή θα δούμε υπουργού εσωτερικών σε κάποια χρόνια να λένε καλύτερα να είχαμε δαπανίσει αυτά τα ποσά κάπου αλλού και όχι στην ανάπτυξη. Και αυτό, δε, και αυτό είναι δικό σας καθήκον να προστατεύσετε την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη και στους στόχους της, δηλαδή τη βιώσιμη εξάλληψη της ε, φτώχειας. Και πραγματικά είναι και αυτή η άποψη που εκφράζω. Είμαστε εδώ όμως για να ε, οριοθετήσουμε τα πράγματα και τις δράσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σεσίλ Κέντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εγώ για την ε, δυνατότητα που μας προσφέρατε να συζητήσουμε σήμερα. Έχω ορισμένες ερωτήσεις και ξεκινώ με την ε, φάση μετά το κοτονού όπου βέβαια ξέρουμε είπατε ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενσωματωθεί στην, ε, μετά το Κοτονού Συμφωνία και η δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ξέρουμε βέβαια ότι η διάσταση κοινοβουλευτική ε, για αυτές τις συμφωνίες ε, στο ισχύουσε και πάνω απ' όλα έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να οπισθοδρομήσουμε, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό που υπάρχει και να το βελτιώσουμε. Ωστόσο δεν είναι σαφές για μένα τι είδους δομή ετοιμάζεται. Έχει συζητηθεί κάποια δομή για την ενίσχυση της κοινοβουλευτική διάσταση ε, και βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε σχέση με τι χώρε ΑΚΕ. Και αυτό το λέω διότι ορισμένες δομές που ήδη υφίστανται το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, παραδείγματι, είναι πολύ αδύναμες και δεν είναι σε θέση να προωθήσουν περισσότερο την κοινοβουλευτική διάσταση. Οι βουλευτές που συμμετέχουν στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο δεν είναι οι ίδιοι που συμμετέχουν ε, στην ε, κοινοβουλευτική συνελευσία και εκπροσωπούν χώρες. Και όχι όλη την Ήπειρο. Ο καθένας στη χώρα του. Αυτά είναι σημεία δυναμίας όμως και πρέπει να αλλάξουν αυτό το πράγμα πλέον. Πάνω απ' όλα δεν πρέπει να πιστοδρομήσουμε και να περάσουμε σε δομές ακόμη πιο αδύναμες από αυτές που επιδιώκουμε. Πρέπει να κάνουμε βήματα πρόοδου, να ενισχύσουμε την ε, δομή την ισομερή δηλαδή κοινοβουλευτική συνέλευση που ήδη υφίσταται μέσα στην οργάνωση του Κοτονού. Λοιπόν, αυτή τη δομή την έχετε αξιολογήσει, τι βλέπετε για την περίοδο μετά το 2020 και επίσης ο Νόρμπερτ Νόιζερ το υπενθύμησε ότι θα πρέπει από τον Οκτώβριο ήδη να έχουμε μια σαφέστερη ιδέα και μερικά ακόμη ερωτήματα σύντομα. Τους τελευταίους μήνες επισκέφθηκα πολλές ε, χώρες, Μαλή, Αιθιοπία, Νότια Αφρική, Νίγηρα, Νιγηρία, ε, για να καταλήξω σε ορισμένα συμπεράσματα, εκ των οποίων τα έξι. Πολλές από τις χώρες για τις οποίες σας ε, ε, μίλησα έχουν πολύ αδύναμες κρατικές δομές και έτσι δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προσεχείς μεγάλες προκλήσεις. Προτεραιότητα λοιπόν δική μας θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση των κρατικών δομών. Γιατί χώρα χωρίς κράτος ούτε προγραμματισμό δεν μπορεί να κάνει. Δεύτερον, για όλες αυτές τις χώρες που έχω επισκεφθεί, εν γέννη, ιδιαιτέρως όμως για τις χώρες που αντιμετωπίσουν κρίση, η κοινωνία των πολιτών δεν υφίσταται. Δεν, έχουμε αρκετή επένδυση, δεν κάνουμε αρκετές επενδύσεις, δεν στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών και αυτό αποτελεί και διάκριση αρνητική, διακριτική μεταχείριση γιατί ε, στερεί ε, η δυνατότητα ε, σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας εκεί να συμμετέχει σε στα κοινά, να ψηφίζει, να εκφράζει γνώμη κτλ. Πρέπει να στηριχθεί λοιπόν και η κοινωνία των πολιτών και δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο να έρθει η ώρα των εκλογών. Πρέπει να ενισχύσουμε την τοπική ε, διακυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και έτσι να καταλάβει ο κάθε πολίτης ότι ανήκει σε μια κοινωνία. Και το άλλο σημείο που έθιξε η συνάδελφος Έλλης Λάιν, ο Νίγηρας, ο οποίος έχει μια, ένα πληθυσμό που αυξάνεται εκθετικά δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει με την πολιτική του την αύξηση της ε, γενετικότητας ε, τα τόσα παιδιά που γεννιούνται καθημερινά. Δεν μπορεί να ανοίγει από ένα σχολείο κάθε εβδομάδα, γιατί κάτι ότι θα χρειαζόταν. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον Ήγηρα, αν και αυτός έχει βληματικό χαρακτήρα, σαν παράδειγμα. Ε, έχοντας μιλήσει λοιπόν με τις αρχές του Νίγηρα, μαθαίνω ότι έχουν βρεθεί σε αδυναμία πλέον να εξασφαλίσουν δομές ε, εκπαίδευση στα σχολεία που έχουν θέσει πια δεν αρκούν για να υποδεχθούν τα παιδιά και τους νέους που γεννιούνται και μεγαλώνουν. Ε, και βλέπουμε ότι κινδυνεύει να αποκλειστεί από την εκπαίδευση μια ολόκληρη γενιά σε όλες αυτές τις χώρες. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε την ε, εταιρική μας σχέση, στην παιδεία και την τον έλεγχο των δημογραφικών τάσεων, γιατί και τη γνωρίζω ότι πολλές φορές προξενεί φόβους αυτή η έννοια, έχει μεγάλη χρησιμότητα γιατί επιτρέπει μια προβλεψιμότητα, προβλέπει να παρακολουθήσουμε με τον έλεγχο των γεννήσεων, που ίσως να, φαίνεται μόνο κατασταλτικός, ε, τι σημαίνει όμως αυτό, τι προσφέρουμε στον πληθυσμό, άμα δεν έχουν τα μέσα οι άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα αυτή καν για να επιζήσουν και κάτι ακόμα για τις γυναίκες ιδιαίτερως. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις για να βγουν οι γυναίκες από την αφάνεια. Σε πολλές χώρες είναι το 70% της οικονομίας, της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά της άτυπης οι γυναίκες. Και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτό το 70% ε, των ε, κοινωνιών, ε, απλώς να μιλούμε για τις γυναίκες και να λέμε είναι σημαντικές οι γυναίκες. Όχι, πρέπει να μπουν σε ένα τυπικό σύστημα, πρέπει να σταματήσει ο αποκλεισμό τους από το σύστημα τώρα για να περάσω στο Κόγκο, την Καμπόν και τον Μπουρούντι, χώρες με μεγάλα προβλήματα σε ανθρωπιστικό επίπεδο, επίπεδο ασφάλειας, και ρωτώ τι είδους συνεργασία και ενίσχυση των πολιτικών μας για την ανάπτυξη σκοπεύουμε να αναπτύξουμε σε σχέση με τις τρεις αυτές χώρες που έχουν όντως τεράστια προβλήματα. Yeah, maybe I could add, add just a few... Ίσως θα μπορούσα να προσθέσω κάτι. Η Τζούλη Σανταρτίνη είπατε μιλήσατε για μια σειρά στρατηγικών για την Ασία, την Ινδία, τη Λατινική Αμερική, δηλαδή για χώρες μεσαίου εισοδήματος, χώρες που δεν είναι, ανήκουν στις ψεχότερες. Υπάρχει μια ανησυχία όμως σχετικά με την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Χτες ε, παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση ε, πώς λεγόταν αυτή η μελέτη που παρουσιάστηκε χτες, ε, αφορούσε ε, τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, η έκθεση Investing in Sustainable Development, τις επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι δεν πάμε καλά σε ό,τι αφορά το στόχο του 0,7% για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας ανακοινώσαμε δεσμεύσεις, θεωρήσαμε ότι η Αφρική είναι ε, προτεραιότητα ε, για την ε, μείωση της φτώχειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αυτοί οι δύο στόχοι είναι ο μόνος τρόπος να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Αφρική. σε κάποιες περιοχές της Αφρικής ε, ξέρουμε ότι θα, έρθουν, θα υπέλθουν κάποιες κρίσεις και αν θέλουμε μια ε, συνολική ε, στρατηγική. Τώρα αυτή τη στιγμή ε, συζητάνε η ε, DG ECO και η DG DEFCO τι συμβαίνει στον Μπουρουντή, σε άλλες χώρες, τι μπορούμε να κάνουμε, με την διπλωματία για να λύσουμε τις συγκρούσεις. Αν δεν κινητοποιηθούμε τώρα όμως για αυτές τις χώρες, φοβάμαι για το τι, θα συμβεί. Χτες είχαμε εκπρόσωπο από το Σουδάν και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε κατάρρευση. Τεράστια κρίση λοιπόν στην Αφρική. Και αν είμαστε σοβαροί, αντί να δημοσιεύουμε εκθέσεις και στρατηγικές, εντάξει, πολύ καλά, αλλά χαρτί είναι. Τι θα γίνει με τα άμεσα προβλήματα Ας ε, σκεφτούμε μαζί πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα άμεσα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ε, των βιώσιμης ανάπτυξης του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει παρουσίαση στον ΙΕ για το πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα συμμετέχουν ευρωβουλευτές γιατί όχι μόνο εκπροσωπούν τους πολίτες, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια. Χωρίς τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα επιτύχουμε τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Και σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, Νομίζω ότι πριν από λίγους μήνες εξετάσαμε πού ε, πανούμε τα χρήματα και είδαμε ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση μειώνονται και το αναφέραμε στην Επιτροπή Εκπαίδευσης. Ναι, βλέπουμε, ναι, ε, υπάρχουν, πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά ε, στην Ουγγάντα μας είπε ένας ε, υπουργός ότι κάποιο παιδί του είπε ότι ουσιαστικά το σχολείο τι είναι, έλεγχος απλώς ενός πλήθους παιδιών. Δεν ε, γίνεται κάτι παραπάνω. Χρειάζονται ε, πρόσβαση στην εκπαίδευση τα ε, παιδιά για να προσαρμοστούν στη ψηφιακή οικονομία. Χρειάζεται κάποιο επίπεδο μόρφωσης, συγκεκριμένες ικανότητες στη σύγχρονη οικονομία. Χρειάζονται λοιπόν δράσεις υπέρ της εκπαίδευσης. Έχουμε πολλή δουλειά και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μόνο άμεσες βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες. Χρειάζονται χρόνια για να λυθούν κάποια προβλήματα. Ε, και στις δικές μας χώρες χρειάζονται 20-30 χρόνια για να ε, προωθήσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη και για καλύτερη κατανομή του πλούτου. Ελπίζω λοιπόν και στο μέλλον να έχετε, συνεχίσετε να εστιάζετε στην εξάλληψη της φτώχειας. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και για τις παρατηρήσεις σας και για τις ε, για το προσανατολισμό που δίνεται σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το νέο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τομεακές προτάσεις που θα καθορίσουν πολλές δράσεις στο τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό που ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει και αυτό που καταφέραμε στην πρότασή μας για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η εξωτερική δράση και η συνεργασία για την ανάπτυξη να ανήκουν στους τομείς όπου είναι απαραίτητη η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο όχι να μειώσουμε τη χρηματοδοτική ικανότητα, αλλά να την αυξήσουμε στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η συνεργασία για την ανάπτυξη, λοιπόν, θα ανήκει στις πολιτικές που θα χρηματοδοτεί και θα αποδείξουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετική θέση στο τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και στο τομέα της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο μέλλον. Και τώρα πρέπει να εξετάσουμε τη δομή και την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε σε ό,τι αφορά τις ε, ε, δράσεις και τις ικανότητες χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ο διαρθρωμένος διάλογος σήμερα είναι μια καλή εισαγωγή για τον καθορισμό των ε, ευρωπαϊκών μέσων και μηχανισμών για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτά τα ζητήματα όταν θα έχει ε, δημοσιευθεί η πρόταση και ε, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σήμερα όμως ε, εξετάσουμε και κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα και θα είναι σημαντικά ε, για το νέο ε, πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων. Χρειάζονται, χρειάζεται ξεκάθαρος προσανατολισμός στο τομέα της ανάπτυξης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για καθοριστικό στόχο και σημαντική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής. Συμφωνώ ότι πρέπει να προσαρμόσουμε ε, τις ικανότητές μας, τα μέσα μας, προκειμένου να επιτρέψουμε το στόχο, το σημαντικότατο στόχο της εξάλληψης της φτώχειας. Φυσικά δεν είναι καθορισμένο το πώς θα επιτύχουμε την εξάλληψη της φτώχειας. Πρέπει να ε, οικοδομήσουμε τη δράση μας ε, ε, μαζί ε, σε αυτή την πορεία προς την επίτευξη του στόχου της εξάλληψης ε, ε, της φτώχειας στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπου η ανάπτυξη είναι ένας ευάλωτος τομέας και σε ό,τι αφορά τα γεωγραφικά κριτήρια πρέπει να εστιάσουμε στην Αφρική και πιο συγκεκριμένα, ε, και πιο συγκεκριμένα στην υποσαχάρια Αφρική στις αναπτυξιακές μας δράσεις ό,τι αφορά το στόχο του 0,7 του εθνικού ακαθάριστου εισοδήματος είναι πολύ σημαντικός ε, στόχος όταν βλέπουμε την πορεία και την πρόοδο βλέπουμε ότι όλοι μαζί, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου, πολύ ε, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το στόχο του 0,7% του ε, καθάριστου εθνικού εισοδήματος ε, για την βοήθεια στις λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες και για την εξάλληψη της φτώχειας σε αυτές τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των δράσεων, τη λεγόμενη ε, και αυτό το ζήτημα είναι εξίσου σημαντικό. Θα ήθελα πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα το 95 96% των δράσεων του ε, σημερινού ε, προϋπολογισμού είναι συμβατό με την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και όλα τα νέα μέσα και η πρόταση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ως στόχο να διατηρηθεί αυτή η δομή της εξωτερικής μας δράσης. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στην εξωτερική δράση που θα καθοριστούν ακόμα καλύτερα ως τομείς που δεν ανήκουν στην αναπτυξιακή συνεργασία ή στην εξωτερική δράση και στη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων ή ακόμα οι δράσεις που αφορούν τη σταθερότητα και την ειρήνη ε, ε, στα πλαίσια του μηχανισμού για την Αφρική. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτές οι δράσεις θα αποκλειστούν από τον προϋπολογισμό και ε, θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό μέσο χρηματοδότησης, κάτι που συμβάλλει στο να διατηρήσουμε τη χρηματοδότηση των κύριων δράσεων της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρετε σήμερα, όπως η ευελιξία του νέου χρηματοδοτικού μέσου, το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διάφορες δράσεις και το πώς θα υλοποιηθεί το ε, χρηματοδοτικό αυτό ε, μέσο και τα διάθετα ποσά που θα ε, χρησιμοποιηθούν. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να συζητηθούν στο μέλλον να τα συζητήσουμε μαζί και να ε, προσπαθήσουμε να τετραγωνίσουμε το κύκλο, όπως είπατε πολύ σωστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις, κάποιες από τις παρατηρήσεις επικεντρώθηκαν στο θέμα της ε, συνεκτικότητας στο τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και πρόκειται ε, για σημαντική συμβολή της ε, νέας ε, δομής του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η ενίσχυση της αναπτυξιακής πολιτικής, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί περισσότερη συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα ε, τι επιτυχάνει κάθε πολιτική και την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και οι στόχοι αυτοί κάποιες φορές ε, ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής είναι αντιφατικοί με, αυτού, με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως ε, είπατε προηγουμένως, μιλήσατε για, τους στόχους, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για το ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων σε κάποιες ε, περιοχές. Άρα πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα για μας και είναι σημαντικό να καθορίσουμε μαζί και να ενισχύσουμε την ε, ε, συνοχή των διαφόρων πολιτικών. Θα συντάξουμε μια έκθεση που θα δημοσιευτεί τον Ιούλιο του 2019 με στόχο να παρουσιάσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και εντός των συνόρων της και εκτός. Και όντως πρόκειται για έναν ακόμη τομέα όπου η συμβολή μας και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία και στην παρουσίαση αυτής της έκθεσης είναι ε, πρωταρχικής σημασίας. Η σημερινή συζήτηση είναι πραγματικά πολύ σημαντική για την επόμενη φάση των συζητήσεων, διαπραγματεύσεων για το νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας ε, ε, τις γνώμες που εκφράζονται στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που μας ε, κάνατε μια περιγραφή του τι ισχύει. Δεν θα καμφθούμε, θα συγκινήσουμε τις γραφειές μας και πάλι σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα και σίγουρα πρόκειται να ε, έρθουμε σε επαφή με τους συναδελφούς των συναρμοδίων επιτροπών εδώ στο Κοινοβούλιο και βέβαια περιμένουμε να ξανέρθετε να μας παρουσιάσετε το νέο πρόγραμμα των αυτοδημιουργών μετά τον Ιούνιο και πάλι ευχαριστούμε.